Επόμενο θέμα είναι η προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Ξεκινάμε με νέους συμμετέχοντες στη συζήτηση, οπότε να σας επενθυμίσω ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη χρονική πίεση απόψε και παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο αγόρευσης. Στρέφουμε πρώτα προς τον κύριο Χάρμπορ που συνέταξε το ερώτημα και έχει το, την ερώτηση συγγνώμη και έχει το λόγο για πέντε λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, είναι προνόμιο για μένα να μπορώ να κάνω την πρώτη παρέμβασή μου στην αίθουσα από όταν εξελέγει πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και να παρουσιάσω αυτό το θέμα εκ μέρους όλων των πολιτικών ομάδων της Επιτροπής και των συντονιστών και χαίρομαι που πολλά νέα μέλη της Επιτροπής είναι εδώ να με υποστηρίξουν και να συμβάλλουν στη συζήτηση. Δεν νομίζω ότι το Κοινοβούλιο χρειάζεται ε, να του υπενθυμίσουμε τη σημασία που έχει η οδηγία περί υπηρεσιών. Ε, ε, θέλουμε να απελευθερώσουμε την δύσχη τη εσωτερική αγορά σε έναν τομέα που εκπροσωπεί το 70% πιθανότητα τη ευρωπαϊκή οικονομία. Θα δημιουργήσει θέσει απασχόληση και θα έχει δυναμικέ συνέπειε. Και είναι πράγματα που τα χρειαζόμαστε πάρα πολύ, διότι αντιμετωπίζουμε αποτελμάτωση οικονομική. Είναι πολύ ευρύ οδηγία, καλύπτει πολλά έχει πολλά νέα χαρακτηριστικά, είναι περίπλοκη σε πολλού τομεί. χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο με συνεπή και πλήρη τρόπο είναι ζωτική σημασία για να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Στο επίκεντρο της οδηγία είναι το εξή γεγονό. Τα κράτη-μέλη θα άρουν φραγμού για τι επιχειρήσει και πιο συγκεκριμένα μέτρα στην εθνική του νομοθεσία που δημιουργούν διακρίσεις κατά υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες και θέλουν να λειτουργήσουν. Και πιστέψτε μου, υπάρχουν εκατοντάδες νομοθετικές προτάσεις, εκατοντάδες νομοσχέδια και νομοθετήματα σε διάφορα κράτη-μέλη πρέπει να τροποποιηθούν λόγω αυτής της προτάσεως. Εκτός αν όλοι οι συνάδελφοι κινηθούν όλοι μαζί και όλες οι χώρες κινηθούν να το πετύχουν αυτό, αυτή η διακρίση θα εξακολουθεί να παραμένει. Αυτό θα πρέπει να γίνει με συνέπεια. Διαφορετικά αυτοί οι φραγμοί θα παραμείνουν. Και γι' αυτό θέλω καταρχάς να ποτίσω φόρο τιμής ιδιαίτερα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ηγήθηκε όσον αφορά το συντονισμό της όλης διαδικασίας ε, για να εφαρμόσουν την ομοθέσια τα κράτη-μέλη. Και να ευχαριστήσω το Συμβούλιο και τα επόμενα Συμβούλια από όταν υιοθετήθηκε αυτή η οδηγία του 2006 που ηγήθηκαν της διαδικασίας και το είδαμε αυτό σε συνόδους κορυφής που ζητούσαν τη συνεχή εφαρμογή ευσοδηγίε και σωμάτου εθνικά δίκαια. Προ Σεσίλια Μάλστρομ που είναι εδώ, θέλω να πω ιδιαίτερω πώ εντυπωσιάστηκε η Επιτροπή με τη δουλειά που κάνει η Σουηδία όταν πήγαμε στη Σουηδία σε μια αποστολή το Σεπτέμβριο και νομίζω ότι ξεκάθαρα έθεσαν παράδειγμα για πολλού άλλου και πιο ιδιαίτερα ε, ο πολύ προσεκτικό τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζουν το ότι οι δημόσιε αρχέ, όλα τα επίπεδα στη Σουηδία, κατανοούν τι υποχρεώσει που υπέχουν σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο να διοδοτούν εταιρείε που παρέχουν υπηρεσία από άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ανώσεω. Τώρα, το ερώτημά μα απόψε και το ζήτημά μα. Το ερώτημά μας εστιάζεται ιδιαίτερο σε αυτό που θεωρούμε το σημαντικότερο στοιχείο που πρέπει να εφαρμοστεί ταχύτερα δυνατόν. Τα κράτη-μέλη έπρεπε να έχουν μια διαδικασία εξέταση τη νομοθεσία του. Να εξετάσουν ποια είναι τα στοιχεία που οδηγούν σε διακρίσει. Αλλά το Δεκέμβριο, 28 Δεκεμβρίου πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η ενσωμάτωση εθνικά δίκαια για να έρθουν τα εμπόδια. Θα πρέπει μετά οι χώρε όμω να δώσουν κατάλογο με προτάσει όπου πιστεύουν, όπου υπάρχει μένει διάκριση έναντι άλλων χωρών, αλλά δικαιολογείται αυτή η διάκριση προστασία των συμφερόντων της χώρας. Και θα πρέπει οι αρχές των διαφόρων κρατών μελών να εξετάσουν τι κάνουν οι άλλες αρχές άλλων κρατών μελών και να εξετάσουν τις προτάσεις των άλλων εκεί που υπάρχουν διακρίσεις. Είναι μια καλή αφετηρία, μας ενδιαφέρει πολύ. Θέλω να δω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα μας πει, πώς θα προσεγγίσει αυτή η διαδικασία, το Συμβούλιο, τι υποστήριξη παρέχει. επίση θα θέλαμε και κάποια διαβεβαίωση ότι αυτό δεν θα πρόκειται να είναι μια διαδικασία που θα γίνει και κλεισμένων των θυρών διότι οι καταναλωτές και επιχειρήσεις και άλλες ομάδες συμφερόντων θέλουν να γνωρίζουν το πώς εφαρμόζεται η διαδικασία. Θέλουμε να δούμε τον κατάλογο αυτό, θέλουμε να δούμε τον κατάλογο των ρυθμίσεων, των κανονισμών και εσωτερικών καταστατικών που θέλουν να κρατήσουν τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, η ενημέρωση και η πρόσβαση της διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής τεχνολογίας χρειάζεται μια θηρίδα για επαφέ που θα πηγαίνουν, θα απευθύνονται οι επιχειρήσει. Είναι σημαντικό για κάθε ευρωπαϊκή οδηγία. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει αυτέ τι πληροφορίε να τι διαθέτουν, να είναι προσβάσιμε οι πληροφορίε για τι επιχειρήσει, να ξέρουν οι επιχειρήσει τι πρέπει να κάνουν για να μπορούν να κινηθούν και να εμπορεύονται μέσω των συστημάτων. Θα πρέπει να έχουμε πλήρη συστήματα που θα λειτουργούν. Αυτό αφορά, αυτά αφορούν ε, οι ερωτήσεις μας. Θα ήθελα... Ε, ξέρω ότι ο Τσάλι Μακρύβι ο υπεύθυνο και θα το διαβιβάσετε αυτά και δεν μπορείτε να δώσετε πλήρη ενδελεχή απάντηση στην ερώτησή μα. Πρέπει να καταλάβετε όμω και τι προβληματίζει την Επιτροπή μα. Είναι η αφετηρία μια διαδικασία για μα που θα κρατήσει πέντε χρόνια ελέγχου ε, και ασκήσεω πολιτική πίεση επί όλων των κρατών μελών για να συμμορφωθούμε την οδηγία. Απευθυνόμενο προ Σεσίλια Μάστον θα πω ότι απογοητεύτηκα και αυτό είναι λίγο που έχω να πω, ότι ε, την, συζήτησε την έκθεση του Συμβούλιο πέρυσι το Σεπτέμβριο στον φανταγωνιστικότητα. και τι λέει, ότι φαίνεται σε κάποια κράτη-μέλη οι πολιτικές δεσμεύσεις για πλήρη εφαρμογή και έγκαιρη εφαρμογή δυστυχώς δεν έχει υλοποιηθεί. Συνάδελφοι, αυτό δεν αρκεί αυτή η αναφορά. Θέλουμε τα ωφέλη που μπορούμε να αποκομίσουμε και τα θέλουμε τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Χάρμπορ. Καλό που σας βλέπουμε στην Ολομέλεια, στο νέο σας ρόλο και τώρα στρέφομαι καταρχάς προς την κυρία Μάλστρομ, εκ μέρους του Συμβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον Μάλκομ Χάρμπορ και την Επιτροπή Ίντε. Όντως βάζετε ένα πολύ σημαντικό θέμα εδώ. Και η συζήτηση είναι επίση πολύ σημαντική. Όπω είπε και ο Μάικλ Χάρμπορ, η ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών αποτελεί έναν από τον ακρογωνιαίο λίθο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 80% της οικονομίας απασχόλησης, θα αυξηθεί και σίγουρα θα γίνει κάτι όλο και πιο σημαντικό όσο περνάει ο καιρός. Όμως δεν έχουμε δει την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών πλήρως. Πρέπει να φροντίσουμε να έρθουν ό,τι εμπόδια παραμένουν. Δασμών κλπ. Γι' αυτό είναι εξαίρετη ιδέα να υπάρξει αυτή η οδηγία για τις υπηρεσίες και να ενσωματωθεί από τα κράτη-μέλη μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου του έτους. Κάνουμε την τελευταία έκκληση, ώστε όντως να προχωρήσουν τα πράγματα. Πάντως, εκ μέρους του Συμβουλίου θέλω να αναφερθώ σε μερικά ζητήματα βάσει ερωτήσεων που μου έβαλε η Επιτροπή σας. Πρώτα απ' όλα, ο έλεγχος της εθνικής νομοθεσίας σίγουρα βοηθάει ώστε να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό να αρθούν τα τελευταία μέτρα που υπάρχουν για την ελεύθερη κατάσταση, ελεύθερη κυκλοφορία και το κριτήριο της μη διάκρισης. Είναι αναγκαίο. Και η αναλογικότητα επίσης. Αν τα εφαρμόσουμε όλα αυτά, τότε πιστεύω ότι θα μειωθεί και η γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις και τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν το αργότερο 28 Δεκεμβρίου να ε, μεταφέρουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους. Τώρα πολλοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν online υπηρεσίες για να επικοινωνήσουν με τις κυβερνήσεις σε πολλές χώρες. Δεν είναι πάντα εύκολο για όλους, πάντως υπάρχει ένα πιο σύγχρονο σύστημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο μάλλον την επόμενη εβδομάδα η Σουηδική Προεδρία θα έχει μία συνάντηση για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση όπω την ονομάζουμε. Τα κράτη-μέλη στηρίζονται πάντως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γίνονται σεμινάρια για να καταρτιστούν οι αρμόδιοι, να βοηθήσουν ένα τον άλλον με τις καλύτερες, τις βέλτιστες εμπειρίε, Υπάρχει στο σελίδα σε διάφορε γλώσσε και σε γλώσσες εκτός από εκείνη του κράτους μέλους. Όλα αυτά υπάρχουν στην οδηγία. Πάντω οι περισσότερες χώρες, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, θα έχουν πληροφορίες σε πολλές διαφορετικές γλώσσες για τα άτομα επαφής. Έτσι, νομίζω ότι θα υπάρχει αρκετή ενημέρωση ώστε να μπορέσει να αυξηθεί και η προσφορά εργασίας. Τώρα ρωτάτε αν θα τα καταφέρουμε. Θα επανέλθει η Επιτροπή σε αυτό για να πει αν θα γίνει έγκαιρα. Πάντως το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας πιστεύει ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκαιρα. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι ότι ακριβώς η οδηγία είναι συνολική, είναι πλήρης, πηγαίνει πολύ μακριά και δεν πρόκειται μόνο για την νομοθεσία, πρόκειται και για άλλα πράγματα τα οποία βοηθάνε τη συνεργασία. Οι δομέ που θα δημιουργηθούν στα κράτη-μέλη θα κάνουν τη δίκηση πιο σύγχρονη και πιο αποτελεσματική. Βέβαια θα πάρει χρόνο. Ο έλεγχος στη νομοθεσία είναι κάτι τεράστιο, είναι ένα γιγάντιο έργο. Και για να βρεθούν οι λύσεις επίσης διοικήσεις πρέπει να ενημερωθούν για το πώς ακριβώς θα χειριστούν τις αρμοδιότητές τους ηλεκτρονικά και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει σωστή κατάρτιση. Πάντως τα σημεία επαφή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε οι διάφοροι εμπλεκόμενοι να μπορούν να συμμετέχουν και να βοηθήσουν να επικοινωνήσουν προς το κοινό τα θετικά από το νέο σύστημα, αλλά και να πούν ποιες είναι οι ανάγκες τους και οι ανησυχίες τους. Ο διάλογος αυτός είναι κεντρική σημασίας. Οι διάφορες πλευρές έχουν ε, συμμετάσχει μάλιστα και σε δίκτυα όπου αυτά υπάρχουν. Πολλές χώρες έκαναν προτάσεις που το κοινό αντέδρασε για άλλη μια φορά, κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ενδιαφέρον που έχει επιδείξει μέχρι σήμερα για το μέλλον τη οδηγίας αυτή για τι υπηρεσίε. Σίγουρα έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο το Κοινοβούλιο και οι ευρωβουλευτέ, και χαίρομαι που εσεί μα ε, ρωτάτε, ε, θέλετε να μάθετε και εσείς περισσότερα και θέλετε να μάθετε τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Συμφωνούμε για το ότι η οδηγία αυτή που έχουμε πρέπει να εφαρμοστεί έγκαιρα ιδιαίτερα σήμερα που είμαστε σε οικονομική κρίση. Γιατί τα κέντρα αυτά θα βοηθήσουν τον κόσμο και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε και ανάπτυξη και νέες θέσεις απασχόλησης. Ευχαριστώ. Η Επίτροπος. Ε, Κυρία Πρόεδρε, η Προεδρία του, Προεδρία του Συμβουλίου, κύριε Ευρωβουλευτές και κύριε Χάρμπορ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ μέρους του συναδέλφου μου Τσάρλι Μαγκρίβη για όσον αφορά τη συζήτηση αυτή για την οδηγία υπηρεσιών. Δύο, λιγότερο από δύο μήνες πριν από την εφαρμογή της υλοποίησης είναι μια καλή στιγμή για να εξετάσουμε τη δουλειά που έγινε μέχρι τώρα και να αποτιμήσουμε τις εξελίξεις. Η οδηγία περί υπηρεσιών είναι μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες που υιοθετήθηκαν τελευταία χρόνια. Έχει πολλές δυνατότητες να άρει φραγμού όσον αφορά το εμπόριο και την ολοκλήρωση της αγοράς και να εναρμονίσει τις δημόσιες διοικήσεις μας. Και σωστή εφαρμογή γίνεται ακόμα πιο πιεστική ανάγκη στο παρόν οικονομικό πλαίσιο. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα η Επιτροπή ΙΜΚΟ όχι μόνο δραμάτισαν βασικό ρόλο για να υιοθετηθεί η οδηγία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ιδιαίτερα εξετίμησε το συνεχές σας ενδιαφέρον παρακολουθώντας τη δουλειά που κάνουν τα κράτη-μέλη όσον αφορά την εκτέλεση της οδηγίας. Από τη δική μας πλευρά πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε στη δέσμευση που ανέλαβε να διευκολύνει τη διαδικασία εκτελέσεως της οδηγίας. Πήραμε σοβαρά τα αιτήματα των κρατών μελών για τεχνική αρρωγή και καταβάλαμε άνευ προηγουμένου προσπάθειες και πόρους για να υποστηρίξουμε αυτό το έργο. Πάνω από 80 διμερείς συναντήσεις με όλα τα κράτη-μέλη διεξήχθησαν και ομάδες επιρρογνωμόνων συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες πάνω από 30 φορές τα τελευταία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να πραγματοποιήσει την υλοποίηση εθνικό επίπεδο, αυτό είναι ο ρόλος των κρατών μελών και η ενσωμάτωση της οδηγίας υπηρεσιών στο εθνικά δίκαια ήταν μια πρόκληση για τα κράτη-μέλη, ήταν μια πρόκληση διότι συνεπάγεται την υλοποίηση προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας όπως τα σημεία ε, μια ενίας επαφής και απλούστευση νομοθεσίας σχετικά με τις υπηρεσίες. Ήταν κάτι που αντιπροσώπευε πρόκληση διότι συνεπάγεται και εντατικό συντονισμό μεταξύ όλων των επιπέδων των διοικήσεων, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό πώς έχουν τα πράγματα σήμερα και αν θα ανταποκριθούν τα κράτη-μέλη. Πάνω από τα μισά κράτη-μέλη φαίνεται ότι είναι σε θέση να επιτύχουν την εκτέλεση της οδηγίας περιπηρεσιών μέχρι το τέλος του 2009 ή αρχές του 2010. Κάποια κράτη-μέλη ίσως ε, καθυστερήσουν. Αυτό δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικό, κυρίως για πολίτες και επιχειρήσεις που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα δικαιώματά τους στην εσωτερική αγορά παρόλο που η κατάσταση δεν είναι ασυνήθις εν, εν συγκρίση με άλλες οδηγίες εσωτερικής αγοράς, δημιουργεί όμως κάποιες ανησυχίες. Θα πρέπει όμως να λάβουμε επίσης υπόψη ότι ίσως περισσότερο για αυτή από ό,τι για άλλες οδηγίες τα κράτη-μέλη έπρεπε να αντιμετωπίσουν τεράστια τεχνικά, νομικά, πρακτικά προβλήματα. Δοθέντων αυτών το αποτέλεσμα που ελπίζουμε πετύχουμε αρχές του επόμενου έτους ίσως να μπορεί να θεωρηθεί ως αρκετά καλό. Θα ήθελα να απαντήσω λεπτομερέστερα στην ερώτησή σας. Σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη ολοκλήρωσαν τη διαδικασία ελέγχου της εθνικής νομοθεσίας. Κάποια κράτη-μέλη συνεχίζουν την διαδικασία. Ο βαθμός στον οποίο αυτή η διήθηση συνέβαλε σε αποτελεσματική ενσωμάτωση οδηγία στο εθνικό δίκαιο Βέβαια είναι και κάτι δύσκολο να αξιολογηθεί σε αυτή τη φάση. Η προθεσμία είναι στο εθνικό δίκαιο δεν έχει εκπνεύσει ακόμα και τα κράτη-μέλη δεν έχουν υποβάλει ακόμα τι νομοθετικέ αλλαγέ που έχουν επιφέρει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σαφές ότι φιλόδοξη και διεξοδική διαδικασία διήθησης είναι κάτι που χρειάζεται ούτω ώστε να υπάρχει φιλική αντιμετώπιση τη εσωτερική αγορά από πλευρά εθνική νομοθεσία. Και είναι κάτι κρίσιμο και για την ανταγωνιστικότητα του τομέα των υπηρεσιών εν γέννη. Τώρα, όσον αφορά τα σημεία μια επαφή, το ένα σημείο επαφή, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν ένα σημείο επαφής και να έχουν τι δέωσες λύσει για αυτό το σκοπό μέχρι το 2009. Και αυτό δεν θα είναι τέλειο σαν κατάσταση, αλλά πρέπει να αποτελέσει βάση. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξακολουθήσουν ανάπτυξη και αναβάθμιση αυτών των ενιαίων σημείων επαφής που με την πάροδο του χρόνου θα πρέπει να γίνουν κέντρα ηλεκτρονικής εκυβέρνησης. Όσον αφορά αυτό το πλαίσιο, συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό να διατίθενται συμπληρωματικέ πληροφορίε και να υπάρχουν και διαδικασίε που εκτελούνται μέχρι σε αυτών των σημείων αυτών. Κυρίω όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων και την φορολόγηση. Οι επιχειρήσει και οι καταναλωτέ θα πρέπει να γνωρίζουν ποιοι είναι οι εφαρμοστέ οι κανόνε. Όπω γνωρίζετε όμω, αυτό δεν είναι κάτι υποχρεωτικό δυνάμει τη οδηγία. Αναμένουμε, κύριε Πρόεδρε, όσο θα σταθεροποιούνται αυτά τα σημεία μοναδικής επαφή, ενιαίας επαφής και πληροφορίες να αναπτύσσονται. Κάποια κράτη-μέλη ήδη ε, προωθούν το όλο σύστημα. Όσον αφορά τώρα την υλοποίηση της οδηγίας, την εφαρμογή όσον αφορά τις κοινωνικές υπηρεσίες στο βαθμό που καλύπτονται από αυτή την οδηγία, αυτό δεν φαίνεται να έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα. Η οδηγία αυτή καθ' αυτή εμπεριέχει μηχανισμούς που εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες αυτών των υπηρεσιών. Και τέλος, είναι σαφές πιστεύω ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές διαδραμάτισαν ζωτικό ρόλο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής, παρακολούθησαν εκ του σύνεκης προσπάθειες των κρατών μελών και ενεπλάκησαν στην εφαρμογή ποικιλοτρόπως. Και εμείς θα εξασφαλίσουμε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές θα εκφράζουν την άποψή τους του χρόνου κατά τη διάρκεια της αξιολογήσεως των αποτελεσμάτων της εκτελέσεως της οδηγίας. Άρα πρέπει να βρούμε τη μέθοδο με την οποία θα εξασφαλίσουμε ότι αυτή η διαβούλευση θα είναι στοχευμένη και συγκεκριμένη. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, πολλά κράτη-μέλη ε, προέβησαν σαν ανοιχτέ διαβουλεύσεις όσον αφορά το σχέδιο νομοθετημάτων κατά τη διάρκεια τα νομοσχέδια κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων και κάποιοι φορείς ε, διενήργησαν κάποιες, ε, ε, κάποιες έρευνες όσον αφορά την εφαρμογή. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και ειλικρινείς σε αυτό το στάδιο. Πολλά απομένουν να γίνουν στον τομέα της εφαρμογής οδηγίας και τα κράτη-μέλη που έχουν μείνει πίσω θα πρέπει να καταβάλουν και άλλες προσπάθειες. Εγώ είμαι πεπισμένη όμως ότι το ποτήρι το δούμε σαν πάνω από μισογεμάτο αλλά καλύτερα, καλά θα κάνουμε να φροντίσουμε να το γεμίσουμε τελείως και γρήγορα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε, λέει ο Πρόεδρος. Εν τω μεταξύ έχω αναλάβει την ε, ε, Προεδρία της ε, συνεδρίασης και θα ομιλώ ουγγρικά. Ε, ευχαριστώ την κυρία Φερέρο Βάλτνερ και τώρα εν ονόματι των πολιτικών ομάδων δίνω πρώτα το λόγο στον κύριο Σφάμπ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο μας ακούσαμε από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ενθαρρυντικό διότι η Ευρώπη από πλευράς διεθνούς ανταγωνισμού βρίσκεται σε μία θέση όπου πρέπει να τοποθετηθούν σωστά και οι υπηρεσίες και ε, εάν ε, καταφέραμε να καταρτήσουμε αυτή την οδηγία με συμμετοχή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πιστεύω ότι η έκβαση τώρα είναι ενθαρρυντική ε, και ότι το ποτήρι είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο όπως είπε η Επίτροπος. Πρέπει να σας πω ότι ε, δεν έχει μόνο παίξει ρόλο στο παρελθόν το Κοινοβούλιο αλλά θα το πράξει και στο μέλλον. Δηλαδή έχω μία ερώτηση προτού ε, ισχύσει η οδηγία αυτή και να σας ρωτήσω αν έχετε, θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε τη φιλοδοξία να εφαρμοστεί η οδηγία αυτή μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και εάν πρόκειται να καλύψετε τις υποχρεώσεις στους επόμενους μήνες. Εμείς θα παρακολουθούμε εν ονόματι των πολιτών, εν ονόματι των εργαζομένων και στα πλαίσια αυτά θέλουμε να δούμε πώς συμπεριφέρονται τα κράτη-μέλη και τι διαφάνεια υπάρχει σχετικά με την οδηγία αυτή πόσο ελέγχεται, ελέγχεται αποτελεσματικά αν ε, τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις τους προς τους παρόχους ε, υπηρεσιών και στο μέλλον όπως και στο παρελθόν θα παρακολουθούμε πώς ε, εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τη συνθήκη για να μην έχουν εντύπωση οι πολίτες ότι προέχουν τα συμφέροντα των κρατών. Όσον αφορά την ηλεκτρονική διεκπαιρέωση των διαδικασιών, αυτό που είναι σημαντικό για μας πρέπει να δούμε εάν ε, οι υπηρεσιών μπορούν να διεκπεραιώνουν όλες τις διαδικασίες ηλεκτρονικά και ε, ε, εάν τα άτομα αυτά τα οποία κρύβονται πίσω από τις ιστοσελίδες μπορούν να συναντούνται ε, με άλλα άτομα και όχι να κρύβονται πίσω από ένα τείχος. Τέλος κυρίες και κύριοι το Κοινοβούλιο είχε πιέσει να υπάρχει το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης και πληροφόρησης και να γίνει σωστή εφαρμογή της οδηγίας και ελπίζω κυρία Πρόεδρε ότι θα κάνετε ό,τι είναι δυνατόν ώστε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να μπορέσει να ισχύσει αυτή η οδηγία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σβάμπ.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 θα μπορούσατε να είχατε απαντήσει σε μία ερώτηση αλλά καλύψε όλο το χρόνο σας οπότε δεν σας δίνω άλλο χρόνο και τώρα το λόγο έχει η κυρία Γκέπχαρτ ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που ευχαριστώ ιδιαίτερως που συζητάμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και θέλω να πω σαφώς ότι σαν κοινοβούλιο όχι μόνο διαδραματίσαμε ένα ρόλο αλλά φροντίσαμε να υπάρξει ένας λειτουργικός συμβιβασμός σε αυτή την οδηγία παροχής υπηρεσιών και αυτό βασίζεται στα κοινωνικά δικαιώματα και ε, την προάσπιση των κοινωνικών συμφερόντων. Γι' αυτό και χρειάστηκε και όντως υλοποιήθηκε η οδηγία παροχής υπηρεσιών. Ε, βλέπω όμως ότι δεν απαντήσατε στα ερωτήματα τα οποία θέσαμε διότι είναι κρίμα σε αν διαπιστώσουμε ότι ε, ισχύει αυτό που άκουσα από πολλές πλευρές δηλαδή ότι υπάρχουν κράτη-μέλη όπου θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή αυτής της οδηγίας και η ισορροπία την οποία επιτύχαμε για να την τορπιλήσουν και να μην σεβαστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων όπως το έχουμε προβλέψει στην οδηγία αυτή. Και αυτό αναφέρεται σε αμφισβητήσιμες συνθήκες εργασίες και σε ορισμούς οι οποίοι περιγράφονται ή περιορίζονται και όπου σε ορισμένα κράτη-μέλη ε, υπό το πρόσχημα των κοινωνικών υπηρεσιών δεν ε, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις αυτής της οδηγίας. Και θα έλεγα ότι το εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροφής εδώ δεν είναι σωστό διότι μας οδηγεί σε λάθος δρόμο και δεν ακολουθεί τον σωστό ορισμό. Και ήδη αυτά τα παραδείγματα μας αποδεικνύουν ότι χρειάζεται ένα νομικό πλαίσιο για την προάσπιση των συμφερόντων μας κατά τρόπον ώστε ε, το κοινωνικό αυτό δικαίωμα στην εργασία να γίνεται παντού σεβαστό και οτιδήποτε άλλο δεν θα υπαρκούσε. Θέλω, είχα ρωτήσει λοιπόν σχετικά με την εφαρμογή. Έχετε συμβουλευτεί, συμβουλευτεί τους ενδιαφερόμενους ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, έχουν εμπλακεί οι κοινωνικές δυνάμεις. Έχω κάνει αυτό το ερώτημα, δεν έχω ακούσει απάντηση και ευχαρίστω θα άκουγα τι έχετε να μου πείτε από αυτού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κρόιτσμαν είναι ο επόμενος. Κυρίες και κύριοι, η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη γνώμη μου δεν είναι ε, θαρρυντική όπως είπε ο κύριος Σβάμπ, αντιθέτως είναι απογοητευτική γιατί δυστυχώς έχουμε καλύψει το 50% του χρόνου και στο άλλο 50% δεν ε, έχουμε προχωρήσει καθόλου γιατί αν σκεφτώ ότι η Γερμανία ορισμένα κρατήδια έχουν εφαρμόσει την οδηγία και στην δικιά μου πατρίδα ήδη στις 2 Σεπτεμβρίου ε, θα ισχύσει ε, θα έπρεπε να ισχύσει αυτή η οδηγία για τη Ρινανία Φάλτς. Σκεφτείτε τι θα γίνει σε άλλες περιοχές. Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 ζητάτε να υπάρχει μία διαδικασία συνένεση εσείς αλλά αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δεν προχωρά και υπάρχουν δυσκολίες και καθυστερήσεις πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πάρα πολύ δεν πρέπει να υπάρξουν αυτές οι καθυστερήσεις διότι παραδείγματο χάρη ε, πρέπει να δούμε ε, τι θα γίνει με τους ομολόγους μας έχουν τις γλωσσικές γνώσεις γνωρίζουν και έχουν την ε, διοικητική υποδομή να εφαρμόσουν αυτή την οδηγία. Εκεί έχουμε πολλές αμφιβολίες διότι εδώ θα έπρεπε η Επιτροπή να ρωτήσει ποιες χώρες ήδη ε, καλύπτουν, ποιες καλύπτουν αυτό το 50% το θετικό ε, για να ξεκινήσουμε από εκεί ε, και να μην δημιουργηθεί μία καθυστέρηση γιατί είμαι βέβαιος ότι την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους τα περισσότερα κράτη αυτή η οδηγία δεν θα έχει εφαρμοστεί και αυτό είναι πρόβλημα διότι τα κράτη είχαν ήδη τέσσερα χρόνια καιρό. Άρα αυτό είναι πολύ απογοητευτικό. Ευχαριστώ κύριε Κρότσμαν. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Σιμάνσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, στη συζήτηση αυτή θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι έχει γίνει για να βγούμε από την κρίση. Στην Πολωνία, παρά την κρίση και διάφορες άλλες ε, αλλαγές που κάναμε, καταφέραμε να ετοιμάσουμε μία πράξη για τις υπηρεσίες η οποία βασίζεται σε έναν ε, αρκετά μεγάλο βαθμό ελευθερίας στον ε, τομέα επιχειρήσεων που έχουν να κάνουν με ξενοδοχεία, με τουρισμό, με σκάφη αναψυχής ή οτιδήποτε έχει να κάνει με ανταγωνισμό. Ο συμβασμό του 2006 έλεγε ότι οι διάφοροι τομεί δεν θα καλύπτονταν από την οδηγία. Τώρα, τι έχετε να πείτε. Το 2006 είχαμε φανταστεί ότι παρετέρω δουλειά θα γινόταν για τις υπηρεσίες κοινή ωφελία. Τώρα είναι μισοάδιο το ποτήρι και θα έχουμε κι άλλο τέτοιο ποτήρι μισοάδιο. Η κυρία Σβένσον έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, ο συμβασμό τον οποίο καλύψαμε το 2006 ήταν τέτοιο που οι σοσιαλιστέ απέσυραν το αίτημα για κοινωνικέ πτυχέ να συμπεριλαμβάνονται ως προτεραιότητα. Αυτό είναι κάτι που ο κύριος Χάρμπορ δεν έχει υπολογίσει καλά. Ακούσαμε από την Επιτροπή και ήταν ξεκάθαρο ότι όταν υπάρχει διαμάχη μεταξύ διαφορετικών προδιαγραφών αγοράς εργασίας, σε δύο διαφορετικές χώρες δηλαδή, τότε η έδρα της επιχείρησης είναι εκείνη η οποία καθορίζει το πώς θα χειριστούμε μια τέτοια περίπτωση. Υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές που λένε ότι η επιχείρηση η οποία προσφέρει τις υπηρεσίες δεν είναι υποχρεωτικό να έχει μόνιμο εκπρόσωπο στην λόγο χώρα. Οπότε τα συνδικάτα δεν έχουν κανέναν με τον οποίο να διαπραγματευτούν. Οι δικαστικές αποφάσεις θα μπορούσαν να συνεχίζονται όπως είχε ήδη αποφασιστεί. Στη Σουηδία δεν βλέπω άλλο τρόπο να λυθεί το ζήτημα παρά μόνο αν υπάρχει ένα νομικό πρωτόκολλο στις συνθήκες όπου τα συνδικάτα και τα κοινωνικά δικαιώματα θα υπερισχύουν τις ελευθερίες της αγοράς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Τώρα έρχονται οι άλλες ε, ομιλίες και η κυρία Κόμη για δύο λεπτά είναι η πρώτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πάνω απ' όλα η οδηγία των υπηρεσιών αντιπροσωπεύει για την Ευρώπη την τελειοποίηση. Μια διαδρομή της οποίας τελικός προορισμός είναι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για να διευκολυνθεί να διευκολυνθούν οι συναλλαγές εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως και οι διοικήσει μπορούν να συντονίσουν τι προσπάθειε που καταβάλουν και μπορούν να ελαχιστοποιήσουν το κόστο των συναλλαγών μεταξύ των διαφόρων συναλλαγών μεταξύ διαφόρων τομέων στα διάφορα κράτη-μέλη. Εναρμόνιση του περιεχομένου των διαφόρων διοικητικών διαδικασιών και διευκόλυνση τη ελευθερία εγκατάσταση των παρόχων υπηρεσιών σε άλλα κράτη-μέλη σημαίνει αυτομάτως την ανάπτυξη, τόνωση της ανάπτυξης και να το δοθεί ανάπτυξη σε μια περίοδο που περνάμε που είναι ιδιαίτερη κρίση. Η οδηγία των υπηρεσιών που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου του 2006 εντάσσεται πλήρως στο εσωτερικό της στρατηγικής της Λισαβόνας αναθεωρήθηκε και υιοθετήθηκε σε μια συγκυρία σε διάφορες συγκυρίες που πέσει η Ευρώπη την τελευταία εννέα αιτία τελικός στόχος είναι η ευρωπαϊκή οικονομία να γίνει πιο ανταγωνιστική στον κόσμο που βασίζεται όμως σε μια πτυχή της γνώσης, σε μια βάση της γνώσης. Η οικονομική κρίση που περνάμε και που η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σε επίπεδο θεσμικό συντονίζοντα διάφορες παρεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα και στα διάφορα κράτη-μέλη δείχνει ότι έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη σωστής και άμεσης εφαρμογής της οδηγίας των υπηρεσιών κάτι που δεν είχε γίνει τη στιγμή που υθετήθηκε. Η προθεσμία της 28 Δεκεμβρίου του 2009 για την ενσωμάτωση της οδηγίας υπηρεσιών δεν είναι απλώς μια ένδειξη της στιγμής κατά την οποία να αποφασίστηκε να περάσουμε στην επικύρωση μέσω της νομοθετικής διαδικασίας της οδηγίας αυτής, αλλά αντιπροσωπεύει πάνω από όλο ένα σημαντικό βήμα προς μια Ευρώπη που έχει πάντα επίγνωση των μέσων που διαθέτει και που είναι πιο ικανή να εκμεταλλεύεται καλύτερα τους δικούς της πόρους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Βενιό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Η συζήτηση έχει ξεσηκώσει τα πάθη, αλλά μετά η οδηγία αυτή πέρασε χωρίς ε, να τις δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο που πρέπει να σωματωθεί στην Εθνική Νομοθεσία. Το άρθρο 2 αναφέρεται στον αποκλεισμό των κοινωνικών υπηρεσιών από το πεδίο εφαρμογή, όταν πρόκειται για βοήθεια, αρρωγή προς τους έχοντες ανάγκη. Είναι δυνατόν να είμαστε περιοριστικοί στον ορισμό των κοινωνικών υπηρεσιών σε ορισμένε χώρε. Εγώ ανησυχώ πάντω για την ερμηνεία που επίτηδε περιορίζεται και μπορεί να δικαιολογήσει τελικά ε, την συμπερίληψη των ε, περιπτώσεων αυτών στην οδηγία. Οι πολίτες πρέπει να μπορούν να έχουν προστασία. Ελπίζω ορισμένα κράτη, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, δεν θα υποφεληθούν από την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία για να ελευθερώσουν κοινωνικές υπηρεσίες με άλοθη ότι έτσι προσαρμόζονται στην κοινοτική νομοθεσία. Οι υπηρεσίες, οι κοινοφιλείς, μάλλον υπηρεσίες, πρέπει να έχουν ιδιαίτερη ρύθμιση και να μην εξαρτώνται από έναν ε, ορισμό για τις εμπορικές υπηρεσίες. Ε, η επόμενη ομιλήτρια είναι ε, η Γκρέφιν Τούν και Χόχσταϊν. Για δύο λεφτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Προ... Κύριε Πρόεδρε, η σωστή εφαρμογή της οδηγίας υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο για τους Ευρωπαίους επιχειρηματίες που λειτουργούν στην εσωτερική αγορά, αλλά και για τους καταναλωτές. Το παράδειγμα της οδηγίας των υπηρεσιών που, ε, για την οποία διαθέσαμε τρία χρόνια για να υλοποιηθεί έδειξε ότι δεν λειτουργήσε και ότι όχι όλα τα κράτη-μέλη θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν σωστά την οδηγία. Χρειαζόμαστε έξοχο συντονισμό μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και μεταξύ των θεσμών ούτως ώστε να εφαρμοστεί σωστά αυτή σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό έχουμε και τις συστάσεις του Ιουνίου του 2009 για τους τρόπους βελτιώσεως της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Προσωπικά πιστεύω ότι στη διαδικασία εφαρμογής θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Γι' αυτό η έκθεση για το σύστημα βαθμονόμησης εσωτερικής αγοράς οδήγησε την πρόταση για τη δημιουργία ενός φόρουμ για την εσωτερική αγορά που θα παρτίζεται από εκπροσώπους των διαφόρων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, από εκπροσώπους των κρατών μερών και άλλων ενδιαφερομένων μερών, ούτως ώστε να αναλυθούν κάποιες υποχρεώσεις για την εφαρμογή της οδηγίας για να παραχθούν οι αναγκαίες διατάξεις σωστή εφαρμογή της. Είναι πολύ σημαντική αυτή η οδηγία. Θέλω αυτό το φόρουμ εσωτερικής αγοράς να είναι ένας τόπος ανταλλαγής βελτίστων πρακτικών μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως το φόρουμ θέλουμε να εστιάζεται στο πώς λειτουργεί η κοινή αγορά, η ιστορική αγορά. Είμαστε υπεύθυνοι για τη λειτουργία της αγοράς οι πολίτες μας θα πρέπει να συμμετέχουν στην προσπάθεια επίσης. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, αναφερθήκατε εκτενώς σε αυτά, σε αυτή την αίθουσα και γι' αυτό έχω το εξής ερώτημα. Τα κράτη-μέλη ζήτησαν τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν τη αυτή περιπτώσει. Κατάφεραν να εφαρμόσουν κάποιες από τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να βρει νέες λύσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί όλα τα αναγκαία μέσα για να υποστηρίξει τις χώρες εκείνες που αντιμετωπίζουν προβλήματα εκτέλεσης. Εν συντομία υπάρχουν νέες ιδέες επί του θέματος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ ανησυχητικό ότι οι επαφές με την τοπική αυτοδίκηση, τουλάχιστον στη χώρα μου, δείχνουν ότι πολλοί, πολλές τοπικές αυτοδικήσεις δεν γνωρίζουν ακόμα τι τους περιμένει όταν τεθεί σε ισχύ η οδηγία. Πολλοί δεν γνωρίζουν την υφιστάμενη νομοθεσία για τις τέσσερις ελευθερίες. Υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης όσον αφορά τις διατάξεις τους νόμους για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για τις μεταφορές. Υπάρχει πρόβλημα για να προστεύσουν τις διοικητικές διαδικασίες οι διάφορες αρχές και τους κανόνες που ισχύουν για το εμπόριο και την αδειοδότηση. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει περισσότερες πληροφορίες, να βοηθήσει την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές αρχές. Είναι επίσης σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει στη διαδικασία μετά από την εφαρμογή της οδηγίας, αν θέλουμε η εφαρμογή της οδηγίας να αντικατοπτρίζει τα όσα συμφωνήθηκαν στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό ο κύριος Λιμπεράτσχη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ. Σε στιγμές κρίσης πρέπει να προσπαθούμε πιο σκληρά να φτιάχνουμε νέες θέσεις απασχόλησης και να ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Πρέπει επίσης να προσπαθούμε να μειώνουμε τις τιμές γιατί έτσι δημιουργούμε ε, μεγαλύτερη πρόσθετη αξία για άλλα αγαθά. Αυτό λοιπόν που χρειαζόμαστε δεν είναι επιδοτήσεις αυτό που χρειάζεται ο κόσμος είναι θέσεις απασχόλησης. Εγώ έχω ένα παράδειγμα κάποιου φούρνου σε μια γειτονική χώρα και έγιναν επενδύσεις και η τοπική κυβέρνηση τελικά απέσυρε την υποστήριξή της. Γιατί, Γιατί η τοπική οργάνωση ήταν κατά αυτού του νέου φούρνου που είχε κατασταθεί στην περιοχή. Οπότε να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Ποιε χώρε είναι καλέ στην εφαρμογή αυτού του μέτρου και ποιε έχουν μείνει πίσω. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε ξεκάθαρα. Θέλουμε να δούμε πώ εφαρμόζεται συγκεκριμένη η οδηγία αυτή στα διάφορα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε κύριε Λιμπεράτσκι. Κάτσε τι τώρα. Τώρα για πέντε λεπτά θα έχουμε τη διαδικασία Catch the Eye. Ε, έχουν πολλοί ζητήσει το λόγο, θα δώσω όμως το λόγο μόνο σε πέντε. Και πρώτα στην κυρία Χάνλικ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, συμφωνώ με τόσα είπατε για την οδηγία υπηρεσιών για το ότι είναι μια από τις πιο σημαντικές οδηγίες που είχαμε τα τελευταία χρόνια και ότι η εφαρμογή της νομοθετικής αυτής πράξης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στην τελευταία θητεία του Κοινοβουλίου εγώ δούλεψα για την οδηγία αυτή και θυμάμαι τι προσπάθειες έπρεπε να κάνουμε όλοι για να προχωρήσει. Εγώ υποστηρίζω την οδηγία υπηρεσιών, αλλά λέω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για τους επιχειρηματίες και για τις οικονομίες μας, όμως είναι μια ευκαιρία που θα έχει απτά αποτελέσματα εφόσον η οδηγία αυτή έγκαιρα τεθεί σε εφαρμογή στα διάφορα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ με αυτά που είπαν και οι ότι η οδηγία δηλαδή πρέπει να εφαρμοστεί γρήγορα. και να προσέξουμε πάρα πολύ πώς θα εφαρμοστεί στα διάφορα κράτη-μέλη. Στη χώρα μου, στην Πολωνία, η οδηγία αυτή τίθεται σε εφαρμογή αυτή την εποχή και ελπίζω ότι θα έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα σύντομα. Ευχαριστώ. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Χεπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το μοντέλο του σκανδιναβικό τη αγορά εργασία βασίζεται σε συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Αυτού του είδου το μοντέλο δεν θα λειτουργήσει αν κάποιο από του εταίρου, σε αυτή την περίπτωση ο πάροχο υπηρεσιών, δεν έχει κάποιον εκπρόσωπο επιτόπου με τον οποίο μπορεί κανεί να διαπραγματευτεί. Γι' αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερω που ε, ε, ελήφθη απόφαση για την οδηγία περί υπηρεσιών και ελήφθη απόφαση υπό την οποία θα μπορούν να συντάσσονται, να εφαρμόζονται συλλογικέ συμβάσει και θα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Η εφαρμογή της οδηγίας υπηρεσιών στη Σουηδία παρόλα αυτά δημιούργησε συζητήσεις, δηλαδή για το κατά πόσο είναι δυνατόν να επιβάλλει κανείς όρους στις υπηρεσίες που παρέχουν, στις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες. Το ερώτημά μου είναι, κατά κάποιο τρόπο η οδηγία ε, παρεμποδίζει τις φιλοξενούσες χώρες ε, να, να, έχουν κάποιες, να έχουν κάποιον εκπρόσωπο οι εταιρείε που παρέχουν υπηρεσίες ώστε να, να μπορούν να γίνουν διαπραγματεύσει. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Φιγκερέντο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στη συζήτηση αυτή δεν μπορούμε να ξεχνούμε τις σοβαρές επιπτώσεις της εφαρμογής της απελευθερώσεως των υπηρεσιών σε πολλές χώρες όπου ε, όταν ιδίω οι χώρες αυτές είναι πιο αδύναμες και υποφέρουν από την κρίση. Ε, αν στα διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν μπορέσουν να ληφθούν μέτρα τα οποία να προασπίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και ακόμη περισσότερο στο δημόσιο θα έχουμε ακόμη και πιο σοβαρά προβλήματα και ε, θα υπάρξει αύξηση και της φτώχειας και της ανισότητος ιδίως στα άτομα που χρειάζονται περισσότερο βοήθεια και αυτό ισχύει για οικονομικές ε, ομάδες που υπάρχουν και στις πιο πλούσιες χώρες. Ε, άρα η προθεσμία θα πρέπει να γίνει σεβαστή για την εφαρμογή της οδηγίας και θα πρέπει να αξιολογηθούν όλες οι αιτίες ε, αυτής ε, της εφαρμογής. Ευχαριστώ η κυρία Κέλλη. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή ΙΜΚΟ θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ευχαριστειών που τόνισε αυτό το σημαντικό θέμα την εφαρμογή τη οδηγία περιπηρεσιών και κυρίω στα πλαίσια τη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε. Δεν θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουν χώρε ούτε επιχειρηματίε σαν δικαιολογία και επιστροφή στον προστατευτισμό που θα ήταν κάτι καταστροφικό ευρύτερα. Ε, το εμπόριο σε υπηρεσίε μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική ανάκαμψη. η Ιρλανδία πλούτησε από όταν μπήκαμε στο εξωτερικό εμπόριο και η κρίση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα ήταν πολύ χειρότερη στην Ιρλανδία αν δεν είχαμε τη βάση για διεθνέ εμπόριο που διευκολύνεται από την εσωτερική αγορά. Και επίση αν δεν ανοίγαμε τα σύνορά μα στον ξένο ανταγωνισμό. Αυτό δεν είχε, αρνη... είχε αρνητικές συνέπειες για τι εσωτερικέ υπηρεσίε, Αντίθετα, ε, αύξησε τον ανταγωνισμό και την καινοτομία. Αυτό που προτείνεται λοιπόν σήμερα είναι κάτι που υποστηρίζω 100% και τέλος θα ήθελα να πω ότι είναι καλό να ακούμε κάποιον εδώ που λέει κάτι καλό για τον Ιρλανδό Επίτροπο, τον Ζάλη Μακρύβη, που είναι φίλος μου, παρόλο που ανήκουμε σε διαφορετικές πολιτικές ομάδες, πολιτικές οικογένειες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Andres. Η κυρία Άντρες έχει το λόγο. Gracias, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μιλάμε για την οδηγία υπηρεσιών. Η οδηγία αυτή είχε ως αντικείμενο να ενισχύσει την τέταρτη ελευθερία, την ελευθερία της αγοράς. μια που μιλάμε για πετίους, αυτό είναι. Πριν από τρία χρόνια εγκρίθηκε και ορίστηκαν προθεσμίες προκειμένου τα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν τις εθνικές τους νομοθεσίες και να άρουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Πέρασε ο χρόνος και τώρα ήρθε η στιγμή να εκτιμήσουμε, να αξιολογήσουμε την κατάσταση, να δούμε πού βρισκόμαστε. Ρωτάω λοιπόν, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει εναρμόνιση και αν ναι, σκοπεύει να προτείνει κάποια νομοθετική πρωτοβουλία για μια τόσο σημαντική οδηγία όπως είναι αυτή η υπηρεσιών για να αναρμονιστεί η αγορά και τα δικαιώματα των καταναλωτών, των πολιτών και των εργαζομένων. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έτσι κλείνει ο κύκλος των, ε, της διαδικασίας Catch the Eye και δίνω τώρα το λόγο στην Υπουργό κυρία Μάλστρομ ώστε σε πέντε λεπτά να μπορέσει να απαντήσει στις ερωτήσεις οι οποίες εδόθηκαν. Ευχαριστώ που θέσατε αυτό το σημαντικό θέμα. Υπάρχει γενική συμφωνία ότι είναι σημαντική αυτή η οδηγία για τις υπηρεσίες και είναι κατεπήγον να εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατόν η Σουηδική Προεδρία, όπως και προηγούμενες προεδρίες, κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτως ώστε να προχωρήσουν τα πράγματα ομαλά και γρήγορα. Συζητήσαμε σε διάφορα συμβούλια το θέμα, διεξήχθησαν σεμινάρια, διεξήχθησαν συζητήσεις κλπ. Και πράγματι ήταν πάντα στην ημερήσια διάταξη για να ενθαρρύνονται οι διαδικασίες και να προωθούνται όμως παραπομένουν λιγότερο από δύο μήνες, ενάμιση μήνες. Τώρα το θέμα ποιος έχει μείνει πίσω και ποιος όχι μπορεί να αλλάξει. Έχουμε ακόμα χρόνο και στόχος μας και είναι και στόχος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή όλες οι χώρες να εφαρμόσουν την ελογοδηγία μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου. Ίσως να υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις, λυπούμεθα. Ξέρουμε όμως ότι όλες οι χώρες κάνουν ό,τι μπορούν για να κινηθούν γρήγορα και ε, ερώτημα τα σημεία επαφής πώς θα λειτουργήσουν. Δεν ε, υπάρχουν ακόμα. Ο στόχος είναι να λειτουργήσουν ε, με τρόπο φιλικό προς το χρήστη και αποτελεσματικά και να περιέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που απαιτούνται ούτως ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών και οι καταναλωτές να ωφελούνται και τα κράτη-μέλη συνεργάστηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να παράσχουν και φυλάδιο με πληροφορίες που θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες ώστε να διευκολυνθεί το τρόπο η ενημέρωση του καταναλωτή και του πολίτη. Πολλά κράτη-μέλη επίση κάνουν ε, δικέ του προσπάθειες καταβάλουν δικέ για τη διάδοση πληροφοριών περί τη οδηγία. Υπάρχει επίση συμφωνία για κοινό σήμα, λογότυπο για διευκόλυνση των χρηστών να μπορούν να κινούνται ανάμεσα στις ιστοσελίδες και στα σημεία επαφής. κάτι κράτη-μέλη, παρόλο που δεν είναι υποχρεωτικό, θα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων και το εργατικό δίκαιο στα σημεία αυτά επαφής. Η οδηγία των υπηρεσιών δεν εμπεριέχει εργατικό δίκαιο και ε, η απόσπαση εργαζομένων εξαιρείται από αυτό. Απαντώ στο ερώτημα του Σουηδού συναδέλφου. Είναι σουηδικό θέμα το οποίο εξετάζεται και είναι λίγο εκτός, είναι κάπως εκτός της συζητήσεως αυτής θα επανέλθουμε σε εθνικό πλαίσιο στο θέμα. Η οδηγία περί υπηρεσιών είναι σημαντική, θα διευκολύνει τους παρόχους υπηρεσιών, θα διευκολύνει την ελεύθερη ε, μετακίνηση, θα είναι κάτι που θα τονώσει την ανάπτυξη της επενδύσεις, θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και θα είναι σημαντικό για τους πολίτες. Οι πολίτες περιμένουν από εμά αυτό το σύστημα λειτουργεί στο ταχύτερο δυνατόν διότι θα διευκολύνει τη ζωή τους και είναι δική μας ευθύνη να εξασφαλίσουμε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν τόσο ώστε αυτό να συμβεί και θα ευχαριστήσω εκ νέου το Κοινοβούλιο όχι μόνο που συνέβαλε στην λήψη απόφασης για την οδηγία αυτή, αλλά διότι ε, λειτουργήσε σαν φύλακα και πίεζε το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να υλοποιηθεί αυτή η προσπάθεια. Αλλά απομένει κάποιος χρόνος και ενδεχομένω θα επανέλθουμε στη συζήτηση μετά στον επόμενο χρόνο επί Ισπανική Προεδρία, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί το σύνεγγυ ακόμα το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Μάλστρομ, τώρα η κυρία Φεραίρο Βάλτνερ για πέντε λεπτά ε, θα συνοψίσει τη συζήτηση. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, όπως είπαμε και προηγουμένοι, έχουμε, προηγουμένως, έχουμε συζητήσει όλα αυτά τα θέματα έχουμε εξαντλήσει όλα τα θέματα τα οποία αναφερόταν στις διάφορες ιδέες ε, για κοινωνικά και άλλα θέματα. Ε, τώρα πρέπει να ξαναγίνει μεν αυτή η συζήτηση αλλά πρέπει να προσβλέπουμε προς τα κράτη-μέλη για να δούμε αν έχουν ε, εφαρμόσει ή θα εφαρμόσουν. Και βάσει των διαθεσίμων πληροφοριών όπως σας είπα φαίνεται ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών θα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία είτε μέχρι το τέλος του χρόνου είτε στις αρχές του 2010. Άρα τα περισσότερα κράτη τουλάχιστον θα έχουν δώσει το σωστό σήμα και θα είναι σε θέση να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους και τις διοικητικές τους δεσμεύσεις. Αλλά ε, όσον αφορά το νομικό πλαίσιο ε, υπάρχει ε, μία κατάσταση διότι ότι ορισμένες ε, χώρες ε, χρησιμοποίησαν αυτή την αναθεώρηση για απλοποίηση της νομοθεσίας ενώ άλλες χώρες έχουν κάνει μόνο λίγες ε, τροποποίησεις και ε, υπάρχει επίσης ε, το ισχύον ε, ρυθμιστικό πλαίσιο και οργάνωση των κρατών μελών όπου κατά περίπτωση διαφέρει. Όλα αυτά βέβαια εξαρτώνται από το πόσο κάθε κράτος θέλει να απλοποιήσει τις διαδικασίες του. Όσον αφορά την σωστή εφαρμογή, ο συνάδελφος Τσάλι Μακρύβη πολλές φορές έχει τονίσει προ στους, ε, ε, ε, στους εκπροσώπους των κρατών μελών ότι πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία και έχει παρακολουθεί στην εφαρμογή με τις υπηρεσίες τους. Όπως σας είπα έχουν υπάρξει πάνω από 80 συνεδριάσεις διμερείς και οι εμπειρογνώμονες κατά την τριετία έχουν συναντηθεί στις Βρυξέλλες 30 φορές. Είμαστε πάρα πολύ δραστήριοι, παρακολουθούμε συνεργαστούμε τα κράτη-μέλη και όντως ε, προσπαθούμε να προσφέρουμε τεχνική βοήθεια αν το επιθυμούν τα κράτη-μέλη αλλά όπως σας είπα τελικά τα κράτη πρέπει να κάνουν αυτή τη δουλειά και να διαθέσουν τους πόρους. Όσον αφορά την επόμενη χρονιά θα είναι βασικό να διασφαλίσουμε ότι η αμοιβαία αξιολόγηση που προβλέπεται από την οδηγία θα γίνει επικοδομητικά και να αξιολογήσουμε αυξήσουμε την ποιότητα της εφαρμογής, ε, της νομοθεσίας, της λειτουργίας και να έχουμε και αντιδράσεις από τις επιχειρήσεις και τους, ε, τους καταναλωτές. Και τέλος, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και άλλους μηχανισμούς ε, εφαρμογής σε περιπτώσεις παραβιάσεως της νομοθεσίας, αλλά είναι πολύ νωρίς για να αναφερθούμε σε αυτό. Γενικώς όμως θεωρούμε ότι ουσιαστικά οι εργαζόμενοι είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αυτοί ενδιαφέρονται για αυτήν ε, την, ε, ε, την νομοθεσία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο πιο βασικός παράγων, θα υποφεληθούν περισσότερο και ε, ε, προβλήματα τα οποία ε, υπήρχαν λόγω ελήψεως διάφανης νομοθεσίας θα καταργηθούν τώρα μέσω της νέας νομοθεσίας και θα υπάρχει μία πρόοδος διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν γνωρίζει κανέναν ο οποίος προσπαθεί μέσω της εφαρμογής της οδηγίας να μειώσει τα δικαιώματα των εργαζομένων και το λέω σαφώς δεν καλύπτονται τα δικαιώματα των εργαζομένων από αυτή την οδηγία και αυτό ήταν ε, ε, σαφές ή σε το πολιτικό συμβιβασμό μεταξύ του Συμβουλίου των Κρατών Μελών ε, και του Κοινοβουλίου. Άλλωστε σε όλα αυτά τα θέματα το Κοινοβούλιο έχει συνεργαστεί πάρα πολύ στενά και ε, θελήσαμε να σας ενημερώνουμε ε, γι' αυτό και για τον τρόπο εφαρμογής ε, και αυτό πολύ εγκαίρος. Θα παραμείνει ένα βασικό θέμα για να μπορέσει η εσωτερική αγορά να λειτουργήσει καλύτερα και να διαθέσει τις δουλειές τις οποίες χρειαζόμαστε Γι' αυτό και θεωρούμε ότι το πρόβλημα αυτό είναι επίγον, ιδίω λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης. Ευχαριστώ ε, για τα καλά σας λόγια κυρία Επίτροπε οπότε κλείνει αυτό το πρώτο μέρος των ερωτήσεων και ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο μέρος δηλαδή εις ε, τον κοινό προγραμματισμό σχετικά με ε, τις ψυχικές ασθένειες και ιδίως το Αλτσχάιμαρ. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Ρόιλ, ο οποίος έχει καθυστερήσει